συνέπειες έχουν ως προς την παρουσία της ακροδεξιάς στην πολιτική μας ζωή. Βρίσκονται εδώ, είναι ανησυχητικές εξελίξεις και στην Αυστρία και στην Ουγγαρία και πρέπει να δώσουμε ιδιαίτερη προσοχή σε αυτές τις εξελίξεις. Μάλιστα. Με βάση την ημερήσια διάταξη, από τις 11 θα αρχίσουν οι ψηφοφορίες, ε, στις οποίες περιλαμβάνεται και η έκθεση του κυρίου Τόμας Ντόιτς. Επόμενο σημείο στη ημερήσια διάταξη είναι οι μαζικέ θηριωδίε στο γιος της Νιγηρία τον Ιανουάριο και τον Μάρτιο. Εκ μέρου Ευρωπαϊκή Επιτροπή το λόγο έχει ο Επίτροπος Όλι Ρεν. Uh, Πρόεδρε, αξιότιμοι κυρίε και κύριοι βουλευτέ, με πολύ μεγάλη οδύνη ενημερωθήκαμε για τον θάνατο του Μαρομούσα, του πρώην Προέδρου της Νιγηρίας, εχθές το βράδυ, ο οποίος είχε συμβάλει τα μάλα στην, ε, στον εκδημοκρατισμό, στην πολιτική και κοινωνική ζωή στην Νιγηρία, στη σταθεροποίηση, χάρη στις προσπάθειές του, ιδιαίτερος της ε, γενικότερης περιοχής, της υποπεριοχής της Δυτικής Αφρικής. Ο αντιπρόεδρος Κούρλακ ε, αναλαμβάνει τώρα την προεδρία ως αντικαταστάτης του. Θα ορκιστεί από ό,τι ενημερωθήκαμε πολύ σύντομα, ίσως και, μέχρι σήμερα, και, και σήμερα ακόμη. Είναι ο, ο αναπληρωτής του Προέδρου ως ε, ανώτατος δικαστικός και ασφαλώς θα διορίσει αντιπρόεδρο ε, για να είναι η κρατική δομή τέτοια ώστε να μπορέσει να αντιμετωπίσει τα δεινά τη Νιγηρία. Οι συνθήκε που επικρατούν εκεί είναι πολύ ανησυχητικέ. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διαρκώς προσφέρει την υποστήριξή τη όλου αυτού τις Μήνε των ταραχών. Οι βίες συγκρούσει, τόσο στο γιο όσο και στα, στη γύρω περιοχή τον Ιανουάριο και τον Μάρτιο του 2010 κατά τη διάρκεια των οποίων φαίνεται πως εκατοντάδες άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στις θρησκευτικέ και εθνωτικές συγκρούσεις, μας έχουν συγκλονίσει. Είναι χιλιάδες οι άστεγοι που ε, βρίσκουν καταφύγιο σε στρατόπεδα προσφύγων και ιδιαίτερος ε, συμμερίζομαι τις ανησυχίες που εκφράζουν οι κυρίες και κύριοι βουλευτές για τη συνθήκη στην περιοχή του Γιος. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα αντιδράσει αρμοδίως και καταλήλους. Ύστερα λοιπόν από τις εκρήξεις βίας τον Ιανουάριο και Μάρτιο αναπτύξαμε επαφές με τον ε, Ερυθρό Σταυρό που δραστηριοποιείται στην Ιγυρία αλλά και με άλλες τεχνικές οργανώσεις με στόχο πρώτα απ' όλα να αντιμετωπιστούν οι άμεσες ανάγκες των θυμάτων και να περιοριστεί στο μέγιστο δυνατό βαθμό η απώλεια ανθρώπινων ζώων. Επίσης καταγγέλουμε δημοσίως ε, τις εκρήξεις βίας. Η κάθε Άστον, η ε, πρόσωπος ε, των εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης μαζί με, την, με τον κύριο Κουσνέρ, τον κύριο Μίλιμπαντ, εξέφρασε σαφέστατη καταδίκη κάθε μορφής βίας ε, και απεύθυνε έκκληση για την άμεση κατάπαυση των εχθροπραξιών και την αναζήτηση ειρηνικής επίλυσης διαφορές και ε, παραπομπή των υπετίων στη δικαιοσύνη. Το Φεβρουάριο, το Μάρτιο, αντίστοιχα Αντίστοιχες, διαφήματα αναπτύχθηκαν σε επαφή με το ε, Υπουργείο των Οικονομικών της Νιγηρίας ώστε να ελεγχθεί και με οικονομικό τρόπο αυτή η έκρηξη βίας ζητήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση, από, το, από την Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση της Νιγηρίας να διερευνήσει διεξοδικά τις αιτίες των πρόσφατων εκρήξεων βίας και να προσαγάγει τους υπετίου στη δικαιοσύνη του ταχύτερου δυνατό. Μέσα στην τελευταία δεκαετία οι βίες συγκρούσει ε, έχουν προκαλέσει το θάνατο 14.000 πολιτών της Νιγηρίας, έχουν οδηγήσει σε εκτοπισμό 3 εκατομμύρια Νιγηριανών. Και δεν μπορούμε να καταδικάσουμε τους μουσουλμάνους ή να χαρακτηρίσουμε τους μουσουλμάνους ή τους χριστιανούς θύτες ή θύματα, γιατί κατά καιρού υπήρξαν ε, και το ένα και το άλλο αμφότεροι. Δυστυχώς ε, συνήθως πρόκειται για ανθρώπους που βρίσκονται και σε δεινές οικονομικές συνθήκες. Πολλές φορές συγκρούσεις που έχουν ίσως θρησκευτικό υπόβαθρο ουσιαστικά έχουν υποδαβληστεί από έχθρα μεταξύ φυλάρχων, από συμφέροντα ε, περιφερειακά ε, και άλλα. Και η ίσως ε, περιορισμένης εμβέλειας διαφορές μερικές φορές εξελίσσονται και διονγκώνονται σε ματηρές συγκρούσεις. Υποστηρίζουμε λοιπόν τις προσπάθειες για την ανοικοδόμηση της Νιγηρία, ιδιαίτερα μέσω του Διεθνού Σωματικού Ταμείου, με τα προγράμματα ιδιαίτερως για την ειρήνη, την ασφάλεια και την χρηστή διακυβέρνηση και ε, το πρόγραμμα για τη δικαιοσύνη, μέσα από τις ε, συμφωνίε του Κοτονού, αλλά και μέσα από την, ε, τις, τις για την ειρήνη και την κατάπαυση με την Ιγυρία απευθείας. Πιστεύω λοιπόν Πρόεδρε ότι θα πρέπει να ε, επαγρυπνούμε ως προς το ζήτημα των, ε, της ιστορικής έκρηξης βίας στην Ιγυρία. Πρόκειται για ένα ζήτημα το οποίο αξίζει να χαρακτηριστεί ως ζήτημα προτεραιότητα και για την προσεχή υπουργική διάσκεψη των ΗΠΑ Εθνών εφέτος το φθινόπωρο. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε κύριε Επίτροπε. Οι ομιλητές τώρα εκ μέρους της κοινοβουλευτικής τους ομάδας. Και πρώτα απ' όλα εκ μέρους του ΕΛΚ για δύο λεπτά το λόγο έχει ο κύριος Μίτσελ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θέλω κι εγώ να εκφράσω τη συμπαράστασή μου στο λαό της Νιγηρίας μετά από τις πρόσφατες συγκρούσεις και την έκφραση βίας εκεί. Πράγμα το οποίο δείχνει τα ευρύτερα προβλήματα που αντιμετωπίζει η χώρα. Υπάρχει μια ιστορία βίας που είναι πολύ ανησυχητική. Στην πόλη υπάρχουν οι μουσουλμάνοι στο βορρά και οι χριστιανοί στο νότο. Και πολλοί πιστεύουν ότι η βία οφείλεται σε θρησκευτικό μίσος. Χρειάζεται να εξετάσουμε καλύτερα τις αιτίε που προκάλεσαν τις βιότητες αυτές. Έρχομαι από την Ιρλανδία και ξέρω ότι για πολύ καιρό ο κόσμος πίστευε ότι πρόκειται για διαμάχη στην Ιρλανδία μεταξύ καθολικών και προτεστατών. Όμως τα πράγματα δεν είναι τόσο απλά. Υπάρχουν πιο σοβαρά πράγματα, πράγματα που έχουν να κάνουν με τα δικαιώματα των πολιτών. Δεν μπορούμε λοιπόν να μιλάμε απλώς για θρησκευτικό μίσος. Υπάρχουν και κοινωνικοί και πολιτικοί και οικονομικοί παράγοντες που πρέπει να ληφθούν υπόψη πριν καταλήξουμε σε συμπεράσματα για την αιτία της βίας. Επίσης πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι και συγκεκριμένα άτομα οφείλονται και συγκεκριμένες φυλές οφείλονται για τις ε, συγκρούσεις οι οποίες δεν εμφανίστηκαν για πρώτη φορά, έχουν ξεκινήσει από το 2004 και μετά αργότερα το 2007 και 2008. Χρειάζεται διάλογο μεταξύ όλων των πλευρών. Είναι ιδιαίτερα απογοητευτικό ότι χώρα όπω η Νιγηρία, που είναι η 8η χώρα ε, που έχει πετρέλαιο, έχει πληθυσμό που ζει σε ένα μεγάλο βαθμό κάτω από τα όρια, δηλαδή βρίσκεται σε ένδια. Η Νιγηρία λοιπόν πρέπει να μπορέσει να βγει από τη φτώχεια και αυτό θα γίνει με κοινωνική δικαιοσύνη που θα κάνει τον κόσμο να αφήσει τη βία στο παρελθόν και να στραφεί προς την ανάπτυξη. Η Συμφωνία Κοτονού πρέπει να βοηθήσει σε αυτό. Πρέπει να εξετάσουμε λοιπόν τις αιτίε που οδήγησαν στις βιοπραγίες αυτές, στι τυβιοδίε αυτές και να μην επαναληφθούν. Ευχαριστώ. Για 1,5 λεπτό το λόγο έχει ο κύριο Τάις Μπέρμαν εκ μέρου των Σοσιαλιστών. Κύριε Πρόεδρε, φυσικά η ομάδα των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών ενώνει τη φωνή της ε, για την ε, έκφραση συλληπιτηρίων για το θάνατο του πρώην Προέδρου. Τον Ιανουάριο και τον Μάρτιο είχαμε θηριωδίε στο Τζος, κάτι που δείχνει την εκρηκτική κατάσταση, την έκρηθμη κατάσταση που επικρατεί στην περιοχή. Βέβαια, ας μην ξεχνούμε την... και τα άλλα αίτια των ε, ε, διαφορών και των βιοπραγιών που δεν είναι μόνο τα θρησκευτικά αίτια. Η, μεγαλή, η, ευρύτερη περιοχή έχει σπάνι πόρων. Ε, επίσης ε, δεν υπάρχει αρκετή αρρώσιμη γόνιμη γη και αυτή γη γίνεται το μήλο της έρευνας μεταξύ μουσουλμανικών και χριστιανικών ε, κοινοτήτων. Οι κτηνοτρόφοι ψάχνουν απεγνωσμένα για βοσκοτόπους για τα κοπάδια τους. Θα πρέπει να βρούμε έναν τρόπο να σταματήσουν αυτές οι βίες συγκρούσεις και να εξασφαλίσουμε ε, ισότιμες και δίκες ευκαιρίες προς όλους για παιδεία και για εξουσία. Θα πρέπει όλοι αυτοί οι παράγοντες να ληφθούν υπόψη. Ζητούμε δίκαιη και διαφανή δίωξη των αυτούργων των βιοπραγιών. Αλλά δυστυχώς οι τοπικοί άρχοντες απειλούν να προβούν σε, εκτελέσει μόνο και μόνο για να αποφύγουν ε, το συγχρονισμό στις νιγηριανές ε, φυλακές. Οι άνθρωποι περιμένουν χρόνια μέχρι να εκδικαστεί η υπόθεσή τους. Υπάρχουν τεράστια προβλήματα και στην ποινική δικαιοσύνη στην Νιγηρία. Μόνο αν αντιμετωπιστούν και αυτά τα προβλήματα θα μπορούμε να προσβλέπουμε σε δίκη και διαφανή δίκη των αυτούργων των βιοπραγιών. Εκ μέρους των φιλελευθέρων για δύο λεπτά το λόγο κύριο Σαλ Γκέρενς. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πριν από λίγο μάθαμε για, την, για το θάνατο του Μάρου Γιάρα Νταούρ και εκ μέρους της ομάδας μου θα ήθελα να εκφράσω τα συλληπιτήριά μου και την θλίψη μου για τον πρόωρο χαμό του Πρόεδρου της Νιγηρίας. Ο θάνατός του λαμβάνει χώρα σε μια στιγμή που η διαμάχη μεταξύ μουσουλμάνων και χριστιανών λαμβάνει μια κρίσιμη καμπή και μάλιστα ε, οι σφαγές, οι πρόσφατες ε, και θηριωδίες στο Τζος ε, είναι χαρακτηριστικό παράδειγμα και δυστυχώς δεν θα πρέπει να περιμένουμε αυτές τις θηριωδίε για να πούμε ότι υπάρχει στην Ιγυρία ένα μεγάλο πρόβλημα μεταξύ των θρησκευτικών κοινοτήτων. Ούτε μπορούμε γενιαστή φορά, να, λέμε ότι η φτώχεια είναι μία από τι αιτίε των συγκρούσεων ή να διαπιστώνουμε την ανικανότητα των τοπικών αρχών να πατάξουν τη διαφθορά. Θα μπορούσαμε επίση για φορά να μιλούμε για την ε, διαμάχη που υπάρχει για την εξασφάλιση γόνιμων γεών ή των ελάχιστων ε, φυσικών πόρων αυτής της χώρας. Είναι επικαλούμαστε τις κλιματικές αλλαγές που και αυτές συμβάλλουν στην ε, ενίσχυση και διόγκωση των προηγούμενων παραγόντων. Τι θα κάνει όμως η Ευρωπαϊκή Ένωση απέναντι σε αυτές τις συνθήκες. Αναφέραμε το άρθρο 8 της Σύμβασης του Κοτονού για την ενίσχυση του διαλόγου με τις ε, πολιτικές αρχές της χώρας. Θα το κάνουμε. Μπορούμε επίσης να καταδικάσουμε ή να στυλιτεύσουμε τις ε, φρικαλαιότητες και τις θηριωδίες. Το κάνουμε και στο ψηφισμά μας. Ή μπορούμε να εκφράζουμε την αγανάκτησή μας και τη θλίψή μας γιατί αυτή η πλούσια χώρα, πρώτη αφρικανική πετρελοεξαγωγός χώρα, δεν καταφέρνει να επενδύσει τον πλούτο της στην καταπολέμηση της ένδυας. Μπορούμε να τα κάνουμε όλα αυτά, να καταδικάζουμε, να ξανακαταδικάζουμε και να επανακαταδικάζουμε όλη αυτή την κατάσταση, αλλά ελάχιστη ε, ελπίδα υπάρχει να διορθωθεί η κατάσταση. ίδια η Νιγηρία θα πρέπει να πρωτοστατήσει σε μια προσπάθεια ανατροπής αυτής της τάσης και ο, ο Good Luck Jonathan, ο τελών χρέη προέδρου αυτή τη στιγμή, έχει όλες τις αρετές ε, και τις ικανότητες ε, με θαραλέο και αποφασιστικό τρόπο να καταπολεμήσει όλα αυτά τα δεινά της Νιγηρίας. Θα πρέπει να αφήσουμε τη χώρα αυτή μόνη της να σταθεί στα πόδια της και να ευχηθούμε καλό κουράγιο, διάβγεια και την αμέριστη υποστήριξή μας προς αυτόν τον ε, καταπληκτικό άνθρωπο που θα εξασφαλίσει αυτή τη στιγμή την Προεδρία της χώρας. Σας ευχαριστώ κύριε Γκέρλες, εκ μέρους των Πρασίνων για 1,5 λεπτό. Το λόγο έχει η κυρία Κιλ Νίλσεν. Πρόεδρε, η ομάδα των Πρασίνων ε, συμμερίζεται και εκείνη τα συλληπιτήρια που εκφράστηκαν εκ μέρου των συναδέλφων. Υποστηρίζουμε πλήρω το ψήφισμα που αναφέρεται στις ε, φρικαλαιότητε που εκδηλώθηκαν μαζικά στην Ιγυρία, που αποτελεί μόνο όμω ε, ένα μικρό τετραγωνικό του φεού πίνακα που παρουσιάζει η Νιγηρία, γιατί θέλω να μιλήσω ιδιαίτερω για τις φυλακές εκεί, όπου συστηματικά παραβιάζονται ανθρώπινα δικαιώματα. 65% των κρατουμένων στη χώρα αυτή δεν έχουν καταδικαστεί καν από δικαστήριο για οδήποτε έγκλημα. Βρίσκονται κρατούμενοι προφυλακιστέ, περιμένοντα εδώ και 10 χρόνια να δικαστούν. Η Νιγηρία δεν, πρέπει, δεν έχει τίποτα άλλο να κάνει παρά να αναγνωρίσει αυτά τα προβλήματα και να προχωρήσει στις ουσιαστικέ μεταρρυθμίσεις του δικατιστικού του συστήματος. Αλλά ακόμα αυτό δεν έχει συμβεί. Και αναφέρομαι στις φυλακές, διότι η επικαιρότητα, η καυτή επικαιρότητα μας υπενθυμίζει πόσο μικρή αξία έχει η ανθρώπινη ζωή στην Ιγυρία. Πολλό δε μάλλον στις φυλακές. Το Εθνικό Οικονομικό Συμβούλιο της Νιγηρίας ανακοίνωσε το σχέδιό του να εκτελέσει εκατοντάδες θανατοπινητών μόνο και μόνο για να αραιώσει τον πληθυσμό των φύλακων. Μόνο και μόνο γιατί δεν έχει αρκετό χώρο. Τίποτε πιο συγκλονιστικό δεν θα μπορούσαμε να περιμένουμε. Όταν γνωρίζουμε ότι πολλοί από αυτούς τους θανατοπινίτες είναι αθώοι, ότι οι πλούστεροι εξ αυτών δεν είχαν καν τη δυνατότητα σε δίκη ε, ορθή και επίσης ο Υπουργό των Εξωτερικών της Νιγηρίας πριν από ένα διάστημα ε, διακήρυτε ενώπιον των Ηνωμένων Εθνών ότι διατηρούσε ε, de facto moratorium στη θανατική, έναντι της θανατικής ποινής η Νιγηρία τώρα είναι δύσκολο να εξηγήσουμε αυτές τις μαζικές εκτελέσεις που εξαγγέλλονται. Πώς είναι δυνατόν λοιπόν το σύνολο των, δι... των διοικητών της Νιγηρίας να προβαίνει στις αποφάσεις. Για ένα λεπτό εκ μέρους ε, των συντηρητικών και μεταρρυθμιστών, ο κύριος Βαντάλε. Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ. Και η δικιά μου ομάδα στέλνει συλληπιτήρια για το θάνατο του Πρόεδρου της Νιγηρίας. Δεν υπάρχει τρόπος να περιγράψουμε τα τραγικά γεγονότα στο Τζος. Αυτά που έγιναν ήταν πραγματικά τραγικά. Ξέσπασμα βίας, με πολλούς χριστιανούς θύματα. Πρόεδρε, στην ε, Ιγερία πρέπει να λάβει χώρα μια ανεξάρτητη έρευνα για να βρούμε τους υπεύθυνου και να βρεθεί τρόπος να προστατεύονται οι πολίτες. Να προσαχθούν στη δικαιοσύνη οι υπεύθυνοι, γιατί δεν είναι δυνατόν να ανεχόμαστε τέτοια γεγονότα. Έπειτα, από πλευρά των θρησκευτικών ομάδων, να βρεθεί μια λύση με διάλογο μεταξύ τους ώστε να μην επαναληφθούν τέτοια γεγονότα. Πρόεδρε, η Ευρώπη πρέπει να στηρίξει την Ιγυρία, αλλά πρέπει και να την πιέσει συγχρόνως, ώστε αυτό το σπιράλι τη βίας να σταματήσει. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε. Εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Ενωτική Αριστεράς τώρα, το λόγο έχει για δύο λεπτά η κυρία Βερζά. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι. Εννοείται ότι και εγώ εκφράζω συλληπιτήρια προς ε, τον λαό της χώρας για το θάνατο του Πρόεδρου. Εμείς δεν θα υπερψηφίσουμε το κοινό ψήφισμα που σήμερα προτείνεται, διότι πιστεύουμε ότι το ψήφισμα αυτό αντιβαίνει στη δικιά μας ε, άποψη για τις αιτίε που οδήγησαν ε, στις θηριωδίες στη χώρα αυτή. Τις καταδικάζουμε βέβαια και ζητάμε οι υπεύθυνοι να προσαχθούν στη δικαιοσύνη, όμως η Νιγερία είναι μια μεγάλη χώρα που έχει τεράστια παράδοση. Έχει 140 εκατομμύρια κατοίκους. Είναι χώρα πλούσια λέμε εφόσον έχει πετρέλαιο το ΑΕΠ την οδηγεί στη δεύτερη θέση στην Αφρική μεταξύ των αφρικανικών χωρών. Όμως ο περισσότερος κόσμος ζει κάτω από το όριο της φτώχειας. Παρά τον πλούτο που έχει σε πετρέλαιο έχει τεράστιο έλλειμμα. Τι ηρωνία. Δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει τον πλούτο της γιατί δεν μπορεί να επεξεργαστεί το πετρέλαιο. Έτσι λοιπόν η παραγωγή μαύρου χρυσού έχει μειωθεί τα τελευταία χρόνια ακριβώς επειδή δεν μπορεί να έχει τις υποδομές που χρειάζεται για τη δίληση του πετρελαίου. Η Νιγερία, λοιπόν αποτελεί ένα κατάφορο παράδειγμα προσπάθειας διεθνών επιχειρήσεων, με τη συνένεση πολλές φορές δικών μας κυβερνήσεων, να χρησιμοποιήσουν τους πόρους της χώρας αυτής. Μιλάω για πετρελαϊκές εταιρείες και μία μάλιστα από αυτές 40% του ε, Νιγηριανού μαύρου χρυσού. Έτσι λοιπόν οι ανάγκες του κόσμου εκεί βρίσκονται σε δεύτερη μοίρα. Το δέλτα της Νιγηρίας ήταν από τις πιο πλούσιες περιοχές και οικολογικά του κόσμου. Δυστυχώ όμως έχει καταστραφεί και εξαιτία ε, του πετρελαίου και επειδή τοξικά απόβλητα φτάνουν στο χώρο εκεί και αφήνονται. Η Νιγηρία λοιπόν είναι μία από τις χώρες που πλήττεται από την περισσότερη διαφθορά παγκοσμίω. Πολλοί επωφελήθηκαν 325 δισεκατομμύρια από τα 400 δισεκατομμύρια που μπόρεσε να έχει χώρα από το μαύρο χρυσό μπήκανε στις τσέπες διαφόρων ονών από τη Γαλλία και αλλού. Η κατάσταση αυτή είναι απαράδεκτη και το σημερινό ψήφισμα δεν είναι στο ύψος των περιστάσεων. Δεν είναι αυτό που θα έπρεπε να είναι για να δείξει η Ευρωπαϊκή Ένωση την αλληλεγγύη της προς την Αφρικανική αυτή χώρα. Πρόεδρος, ευχαριστούμε. Κυρία Βερζένα, λεπτό τώρα ο κύριος Προβέρα για να μιλήσει εκ μέρους τη Ευρώπης για την ελευθερία και την δημοκρατία. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Ξέρουμε πόσο δύσκολο είναι να εξασφαλιστεί η ειρηνική συνύπαρξη διαφορετικών θρησκευτικών κοινοτήτων, ιδιαίτερω χριστιανών και μουσουλμάνων. Υπενθυμίστηκε πόσο σημαντική, πόσο σοβαρή είναι η κατάσταση. Έχουν χάσει τη ζωή του πάνω από 40.000 άνθρωποι από την ε, επάνωδο στη δημοκρατία του 1999. Δυστυχώ όμως δεν πλήττεται μόνο η Νιγηρία από αυτές τις θρησκευτικέ συγκρούσεις. Και καλό θα ήταν να ε, αναλάβει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο την ε, εκπόνηση ετησίως εκθέσεως για τις συγκρούσεις μεταξύ θρησκευτικών κοινοτήτων ανά τον κόσμο, γιατί νομίζω ότι θα μας δώσει μια πολύ διαφορετική εικόνα για διάφορες χώρες του κόσμου. Και θα ήθελα κύριε Ρένα να ε, σας διορθώσω ως προς αυτό που είπατε ότι η Νιγηρία είναι φτωχή χώρα. Είναι πολύ πλούσια χώρα που δυστυχώς όμως έχει ε, το άχθος να φέρει μια πολύ διεφθαρμένη εξουσία, κρατική εξουσία, θεσμική εξουσία η οποία απομιζά τους πλούτους της. Χρειάζεται λοιπόν να αναπτυχθεί μια νέα ηγετική τάξη η οποία να ακούει τους πόθους του λαού. Ευχαριστώ. Το λόγο έχει ο κύριος Χάνς Πέτερ Μάρτιν, του των εγγεγραμμένων. Η Νιγηρία βρίσκεται στο επίκεντρο της προσοχής πολιτικής μας αλλά και στο επίκεντρο της πολιτικής ενόψη του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος Ποδοσφαίρου που θα διεξαγωγηθεί στην Νότια Αφρική είναι μια χώρα η οποία βρίσκεται σε ένα πεδίο τάσης μεταξύ της επιλογής του κινέζικου δρόμου, της κινέζικης λύσης αν θέλετε, και της ευρωπαϊκής λύσης. Και έχω βαθιά πεποίθηση πως θα πρέπει να την πείσουμε να ακολουθήσει τον ευρωπαϊκό δρόμο και να, να καταγγείλει, να καταπολεμήσει αποτελεσματικά τα ανθρώπιν, τις παραβιάσεις των ανθρώπινων δικαιωμάτων και τη διαφθορά. Στις φυλακές της θα πρέπει, αντί για όλους αυτούς τους αθώους που μένουν προφυλακισμένοι, να βρουν θέση η διεφθαρμένη πολιτική και η διεφθαρμένη ηγετική τάξη. Πρέπει εμείς από την Ευρωπαϊκή Ένωση να υποστηρίξουμε με ισχυρή φωνή τα ανθρώπινα δικαιώματα και να μην μείνουμε μέτοχοι παρατηρητές των παραβιάσεων τους στην Ιγυρία. Ωραία, ολοκληρώσαμε τους εκπροσώπους των ομάδων. Θα περάσουμε στους λοιπούς ομιλητές. Πρώτος ο κύριος Μάουρο για δύο λεπτά. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι, η βία δεν επιλύει τις συγκρούσεις και τις διαμάχες. Αντίθετα, ενισχύει και επιτείνει τις ολέθριες και τραγικές συνέπειές τους. Είναι άδικη, απάνθρωπη η βία και σε καμία περίπτωση δεν είναι κατάλληλο μέσο. Και μάλιστα είναι το λιγότερο αποτελεσματικό μέσο για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που πλήττουν μια ολόκληρη περιοχή. Γιατί τα αίτια των βιοπραγιών μεταξύ μουσουλμανικών και χριστιανικών κοινωνίτων δεν είναι μόνο ο θρησκευτικός, ο ε, θρησκευτικός ε, φονταμενταλισμός, αλλά κυρίως ε, η οικονομική ύφεση και οι οικονομικές διαφορές μεταξύ των εθνωτικών ομάδων. Η Ευρωπαϊκή Ένωση μαζί με την Αφρικανική Ένωση αλλά και την παγκόσμια κοινότητα θα πρέπει να δώσει στην Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση της Νιγηρίας που είναι σε μεγάλο βαθμό υπεύθυνη για την κατάσταση αυτή να καταλάβει ότι για να διευκολυνθεί η ειρηνική συνύπαρξη μεταξύ των κοινοτήτων, των εθνοτήτων και των θρησκειών στη χώρα αυτή, θα πρέπει να κάνει κάτι, γιατί μόνο με τέτοια ειρηνική συνύπαρξη θα βελτιωθεί η κατάσταση σε ολόκληρο το λαό της Νιγηρίας. Και εκτός από τη βελτίωση του συστήματος ε, ανάκρισης διαλεύκασης ε, των ε, εγκλημάτων και της παραπομπής στο δικαιοσύνη των αυτούργων, θα πρέπει να αναλυθεί κάθε απαραίτητη πρωτοβουλία προκειμένου να προωθηθεί ο διαθρησκευτικός και διεθνωτικός ε, διάλογος, αλλά να δημιουργηθεί και μια νέα ηγετική τάξη, όπως ζήτησαν πολλοί. Να διαμορφωθεί μια τέτοια νέα ηγετική τάξη. Και με το ψήφισμά μας θέλουμε να δώσουμε να καταλάβουν ότι μια χώρα που έχει τόσο, τόσο πλούσιο ρηκτό πλούτο και ιδιαίτερα πετρέλαιο, θα έπρεπε να εξασφαλίζει μια καλύτερη όχι μόνο πρόσβαση στους σπόρους αλλά ανακατανομή του φυσικού πλούτου και μάλιστα η συμφωνία της 12 η Δεκεμβρίου 2009 μεταξύ της Νιγηρίας και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής θα μπορούσε να δώσει όθηση προς αυτή την κατεύθυνση. Η ασφάλεια σήμερα βρίσκεται στο επίκεντρο των αναρρύθμιτων προβλημάτων που αντιμετωπίζει η Νιγηρία και η βασική απειλή δεν είναι η ίδια η διαμάχη αλλά οι λόγοι που δημιούργησαν αυτή τη σύγκρουση. Θα πρέπει λοιπόν να, να βοηθήσουμε την Ιγυρία και να την συμπαρασταθούμε προς μια νέα δημοκρατική και κοινωνική ανάπτυξη. Σας ευχαριστώ. Το λόγο έχει η κυρία Κρέτσου. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα και εγώ με τη σειρά μου να στείλω τα συλληπιτήριά μου και τη συμπαράστασή μου προς την Ιγυριανό λαό για το θάνατο του Προέδρου του διαπιστώνουμε ότι προστίθεται στην ίδια κρίσιμη κατάσταση ένας νέος κίνδυνος. Ε, η απώλεια ηγετικών στελεχών εξαιτία της σύγκρουσης. Ε, τα τελευταία χρόνια έχασαν τη ζωή τους χιλιάδες μουσουλμάνοι και ταυτόχρονα και χιλιάδες χριστιανοί. Η παρουσία του στρατού στους δρόμους μπορεί ίσως να σταματήσει τα αντίπεινα της μιας κοινότητας προς την άλλη. Θα πρέπει να διαφυλάξουμε τη δημόσια τάξη για να αποφύγουμε την επανάληψη των θηριωδιών. Ίσως με μια παγκόσμια παρουσία, παρουσία της παγκόσμιας κοινότητας. Θα πρέπει να σταματήσει επιτέλους η ατιμορρησία που χαρακτηρίζει πολλές χώρες της Αφρικής. Θα πρέπει να συλληφθούν οι πέτοι οι εγκληματίε μόνο όταν παραπευθούν στη δικαιοσύνη θα σταματήσουν οι βιοπραγίε. Θα πρέπει όμω αυτό να εμπλακεί και η παγκόσμια κοινότητα, γιατί η διεθνή κοινότητα επικέντρωσε την προσοχή τη στα Βαλκάνια, άρα αμέλησε την Αφρική. Θα πρέπει να στρέψουμε την προσοχή μα και προ την Αφρική. Σα ευχαριστώ, ο Δόκτωρ Τάνοκ, για ένα λεπτό. όταν ήμουν μικρό, θυμάμαι πολύ καλά, να παρακολουθώ στη τηλεόραση εικόνε από τον ε, πόλεμο στην Πιάφρα, στην Ιγυρία φίλιο πόλεμο και δυστυχώς 40 χρόνια αργότερα δεν έχουν αλλάξει και πολλά πράγματα. Στο ΖΟΣ αυτή τη φορά εκατοντάδες ανθρώπων έχασαν τη ζωή τους, σφαγιάστηκαν σε πράξεις ε, βαναυσότητας που μας ε, ε, υπενθυμίζουν ότι η Νιγηρία δεν έχει λύσει ούτε τα προβλήματα τα θρησκευτικά, ούτε τις οικονομικές, κοινωνικές, πολιτικές εντάσεις που τη χαρακτηρίζουν. Και χθε ο θάνατος του Προέδρου, και απευθύνω εδώ τη συλληπιτήριά μου στους Νιγηριανούς, φαίνεται ότι ε, θα ενισχύσει ακόμη περισσότερο τον αγώνα για την εξουσία και την αποσταθεροποίηση στη μεγάλη αυτή αφρικανική χώρα. Γι' αυτό το λόγο και ανησυχώ ιδιαίτερος για το κατά πόσον μπορεί να διατηρήσει την ενότητα της ε, η Νιγηρία. Ο ε, διαβόητος πρόεδρος της Λιβύης Καντάφη έχει απευθύνει ήδη κλήσεις για διχοτόμηση της χώρας αλλά και όχι μόνο αυτός έχουν κληθεί, έχει κληθεί μάλλον η ηγεσία της Νιγηρίας να ε, διχοτομεί στη χώρα μέχρι του χρόνου. Έτσι λοιπόν ε, αποδεικνύεται ότι ίσως τα ποικιοκρατικά σύνορα που έχουν, χαράξει, έχουν χαραχθεί στην Αφρική δεν είναι και τόσο ιερά πλέον. Ευχαριστώ πολύ. Το λόγο έχει ο κύριος Τζο Higgins. Πρόεδρε. Οι σφαγές στην Ιγυρία τον Ιανουάριο και το Μάρτιο προκάλεσαν πολλά θύματα και κυρίως γυναίκες και παιδιά. Θρησκευτικές, φιλετικές διαφορές έχουν προκαλέσει πολλές άλλες φαγές και εγκλήματα. Πρέπει όμως να κοιτάξουμε τους ε, βαθύτερους λόγους αυτών των ε, εντάσεων. Το απεικιοκρατικό παρελθόν που χαρακτηρίζει ακόμη και έχει αφήσει βαθιά στίγματα στην Αφρική ολόκληρη η βαριά αυτή κληρονομιά που άλλωστε χαρακτήρισε και το BBC νωρίτερα με μια ανάλυση του στις ε, συνθήκες φτώχειας που αντιμετωπίζουν μαζικά οι Νιγηριανοί και την τεράστια διαφθορά που χαρακτηρίζει την ηγετική του τάξη και που οδηγούν τελικά σε θρησκευτικέ συγκρούσει μεταξύ των φτωχών που είναι και οι μουσουλμάνοι και οι χριστιανοί. Παρά το πολύ πετρέλαιο που διαθέτει η Νιγηρία Δυστυχώς όμως η διεφθαρμένη εξουσία και οι πετρελαϊκές εταιρείες με πρώτη τη Shell απομίζουν το μεγαλύτερο μέρος του πλούτου της χώρας και αφήνουν σε εξαθλίωση και φτώχεια τον πληθυσμό της. Στέκω λοιπόν στο πλευρό του σοσιαλιστικού κινήματος της Νιγηρίας που απαιτεί με τους αγώνες του να επανεθνικοποιηθεί ο πλούτος και να διατεθεί, να αναδιανεμηθεί μεταξύ των πολιτών της χώρας. Χωρίς τον πλούτο αυτό δεν θα μπορέσει να ανοικοδομήσει η Νιγηρία τη ζωή της, δεν θα μπορέσει να εξασφαλιστεί ζωή αξιοπρεπής για τους Νιγηριανούς ή να κλείσουν τα χάσματα και οι πληγές του διχασμού. Η άλλη λύση, που θα, η άλλη εναλλακτική θα ήταν η διχοτόμηση και η συνέχιση των βαρφαροτήτων και βιοπραγιών εις βάρος των αθώων. 1,5 λεπτό παρακαλώ για τον κύριο Κατσμάρεκ. Κύριε Πρόεδρε, κυρίε και κύριοι, η Νιγηρία είναι πάρα πολύ σημαντική χώρα, γι' αυτό και ασχολούμαστε με τα συμβάντα της 7 η ε, Μαρτίου στην περιοχή Τζος. Το πρόβλημα της Νιγηρίας δεν έγκυται στο ότι έχασαν τη ζωή τους χριστιανοί, γιατί τον Ιανουάριο, τον προηγούμενο Ιανουάριο έχασαν τη ζωή τους και μουσουλμάνοι. Εκτός από τις θρησκευτικέ διαμάχες και διαφορές υπάρχουν και άλλες διαφορές, εθνοτικέ, οικονομικές, κοινωνικές, αλλά και δύο άλλα είδη διαφορών, ιστορικέ διαφορέ, γιατί η οι χριστιανοί θεωρούνται ως αυτόχθονες, ενώ οι μουσουλμάνοι ως αλλοδαποί, ως άνθρωποι που ήρθαν τις τελευταίες γενιές μόνο. Υπάρχουν και πολιτικές διαφορές, γιατί οι χριστιανοί ε, είναι, ανήκουν σε ένα κόμμα, ενώ οι μουσουλμάνοι ανήκουν στην αντιπολίτευση. Υπάρχουν τεράστιες διαφορές και δεν είναι μόνο θρησκευτικές διαμάχες οι βασικές συγκρούσεις στην Ιγυρία. Το Σύνταγμα της Ιγυρίας κατοχυρώνει την ανεξιθρησκεία, την ελευθερία της θρησκευτικής λατρείας και την δυνατότητα προσιλητισμού σε άλλη θρησκεία. Είναι κάπως περίεργο και μάλιστα οι αξίες που κατοχυρώνονται σε ένα από τα παλιότερα συντάγματα, το αμερικανικό και στη, το πολωνικό που είναι από τα χειρότερα της ε, ε, Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι τα πιο σημαντικά. Θα πρέπει να καλέσουμε τις ε, αρχές της Νιγηρίας να επιλύσουν αυτά τα προβλήματα, όχι μόνο να προσετερήσουν τις δικές μας αρχές, αλλά να διορθώσουν την κατάσταση στην Νιγηρία. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, πολύ σημαντικό το Σύνταγμα και πολύ σημαντικό και το ψήφισμά μας. Σας ευχαριστώ με τον κύριο Κασμάρικ τέλειωσε ο γύρος των ε, ομιλητών. Περνάμε στο Catch the Eye. Η κυρία Αντρικενέ είναι η πρώτη. Πρόεδρε, θέλω να εκφράσω τη θλίψη μου για την ε, βία που έχει ξεσπάσει στην περιοχή του Τζος με αποτέλεσμα το θάνατο εκατοντάδων ε, ανθρώπων. Είναι πολύ σημαντικό να υπάρξει μια διαδικασία συμφιλίωσης η οποία να βοηθήσει σε ειρηνική συνύπαρξη των ε, μουσουλμάνων και των χριστιανών. Οι βιοπραγίες έλαβαν χώρα κυρίως εξαιτίας της στόχιας, εξαιτίας της καταπίεσης των κατοίκων που ζουν στις πιο φτωχές περιοχές που δεν μπορούν να υποφεληθούν από την ανάπτυξη στη χώρα. Οι αρχές της χώρας λοιπόν πρέπει να φροντίσουν για μια πιο καλή κατανομή του πλούτου για δημοκρατικές αξίες, για ανθρώπινα δικαιώματα. Τέλος, κυρίως σήμερα θέλω να εκφράσω τη συμπαράστασή μου στο λαό της Νιγηρίας για την απώλεια για το θάνατο του πρόεδρου τους. Ευχαριστούμε κύριο Πρέδεκ, τώρα το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θέλω και εγώ να εκφράσω τα συλληπιτήριά μου στο λαό της Νιγηρίας μετά το θάνατο του Πρόεδρου τους, του Γιάρ Αντουά. Θέλω να αναφερθώ πιο συγκεκριμένα σε δύο στοιχεία. Πρώτα απ' όλα, θέλω να ξεκινήσω από κάτι που είπε ένας κάτοικος της Νιγηρίας, τον ρώτησαν τι φταίει για όλα αυτά τα δεινά της χώρας του. Είπε λοιπόν εκείνος ότι οι υπεύθυνοι των ε, θηριωδιών που έλαβαν χώρα εκεί να διωχθούν. Και όχι όπως γίνεται τώρα να εξαφανίζονται. Ποτέ δεν βρίσκονται υπεύθυνοι και δεν διώκονται τελικά. Η μορισία λοιπόν φταίει. Έπειτα δεν πρέπει να ξεχνάμε και τη θρησκευτική διάσταση πολύ πριν από μένα εδώ είπαν ότι υπάρχουν βέβαια θρησκευτικέ διαφορές, αλλά η ουσία του προβλήματος είναι κυρίω οικονομική και κοινωνική. Ο πρόεδρος Goodluck Jonathan το λαμβάνει αυτό υπόψη και γι' αυτό και ζήτησε να έρθουν οι ηγέτε στη χώρα για να συζητήσουν. Ο κύριο Ζήπτορ είναι επόμενο. Ευχαριστώ. Οι εικόνες ε, που είδαμε πρόσφατα σε διάφορες ε, τηλεοπτικές ειδήσει ήταν ανατριχιαστικές και συγκλονιστικές. Είχαμε δολοφονίες ε, εκατοντάδες ανθρώπων στο Τζος. Οι θηριωδείς αυτές πραγματικά μας συγκλώνησαν. Όπως είπε ο συνάδελφος Μάριο Μάουρο, δεν μπορούμε να δικαιολογούμε τη βία. Η βία είναι ούτως ή άλλως κακή. Και η Ευρωπαϊκή Ένωση και εμείς τους Ευρωβουλευτές δεν μπορούμε να αγνοήσουμε αυτό το θέμα. Γι' αυτό και πολύ θερμά υποστηρίζω το ψήφισμα αυτό. Θα πρέπει να δούμε τα αίτια ε, που είναι πολυσχεδή και πολύπλευρα και που οδήγησαν σε μια σειρά συγκρούσεων που δεν είναι μόνο θρησκευτικέ. Τα θέματα δημοσίων ελευθεριών και τα δικαιώματα, τα θεμελιώδη δικαιώματα του ανθρώπου θα πρέπει να γίνουν σεβαστά και στην Ιγυρία. Θα ήθελα να στείλω τα συλληπιτήριά μου προς τον Ιγυριανό λαό για, για το θάνατο του Προέδρου της Ιγυρίας. Θα ολοκληρώσει τη συζήτηση ο Επίτροπος Όλη Ρεν, απαντώντας ε, στα διάφορα σχόλια. <clears throat> Uh, uh, Πρόεδρε, ξέρετε κύριε και κύριοι. Ευχαριστώ για την ε, πολύ σοβαρή και υπεύθυνη συζήτηση που αναπτυχθήκε σήμερα. Πολύ εξημών υπογραμμίσατε το ε, πόσο περίπλοκα είναι τα, προβλήματα, τα κοινωνικά προβλήματα που γνωρίζει η Νιγηρία. Συμφωνώ μαζί σας η Επιτροπή είναι εν γνώση του πλέγματος προβλημάτων που χαρακτηρίζουν τη χώρα. Είμαστε πάντα στο πλευρό της Νιγηρίας, εταίροι και δεν μπορώ παρά να συμφωνήσω μαζί σας ότι είναι άκρο σημαντικό να καταπολεμηθεί η διαφθορά και η ατιμορρησία. Δυστυχώς η διαφθορά έχει βαθιές ρίζες στην Νιγηρία και παρεμποδίζει την κοινωνική πρόοδο και τον εκδημοκρατισμό στη χώρα αυτή που έχει τόσο πλούσιους πόρους. Έτσι οι χαμένοι είναι πάντα οι απλοί πολίτες. Έτσι λοιπόν θα πρέπει να αναπτυχθεί μια σειρά, να αξιοποιηθεί μια σειρά μέσων, διπλωματικά μέσα, αναπτυξιακή βοήθεια, και η Επιτροπή με μεγάλη προσοχή παρακολουθεί τις εξελίξεις με στόχο να συγκρατήσει την έξαρση της βίας στη χώρα αυτή. Το επόμενο, η επόμενη διεθνής διάσκεψη που θα ασχοληθεί με το σημαντικό αυτό θέμα σε υψηλό επίπεδο είναι η προσεχής υπουργική διάσκεψη Ευρωπαϊκής Ένωσης Νιγηρίας στο Φθενόπορο και βεβαίως θα επισημάνουμε όλα αυτά τα ζητήματα επί τη ευκαιρία αυτή. Ευχαριστούμε πολύ και ζητώ συγγνώμη για την φασαρία που ακούγεται στην αίθουσα. Υπάρχουν 7 προτάσεις ψηφίσματος για να κλείσει η συζήτηση αυτή. Η ψηφοφορία θα λάβει η χώρα σήμερα από τις 11 και μετά. Διακόπτουμε για ένα λεπτό προκειμένου να μπορέσουμε να ξεκινήσουμε τις ψηφοφορίες σε λίγα λεπτά.